Πέντε φίλοι, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια μακροσκελή ψηφοφορία ενωπιών μας. Σας παρακαλώ να είμαστε οργανωμένοι, γιατί θα έχουμε τουλάχιστον 2,5 ώρες ψηφοφοριών. Πριν ε, τις διακοπές βέβαια μπορούμε να το κάνουμε για να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας. Επιτυχώς. Λοιπόν, να ξανακάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία, γιατί κάποιοι άλλαξατε θέση. Πρέπει να ξαναλέξουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πιέστε το κουμπί. Άρχεται η ψηφοφορία. Hey. Please vote. Ψηφίστε παρακαλώ. And I close the vote. Λήξη. Νομίζω λειτουργεί το σύστημα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τις εκθέσεις. Καταρχήν, πράξη για την ασφάλεια στον κυβέρνο χώρο. Η κυρία Νίμπλερ είναι η συγγετρία. Θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, στις πολιτικές ομάδες για την υποστήριξη και την καλή συνεργασία που είχαμε εδώ και μήνες. Ε, εργαστήκαμε σκληρά για τους συμβιβασμούς ε, και θέλω να ευχαριστήσω και τη γραμματεία, χωρίς τη γραμματεία που μας συνόδευσε στην προσπάθεια επίτευξη συμβιβασμού, δεν θα είχαμε πετύχει. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σε αυτό το πολύ σημαντικό φάκελο και ενυπομονώ για ένα καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι χωρίς τη γραμματεία δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Συμφωνώ μαζί σας, λοιπόν, 100%. Σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Λοιπόν, λιμπένα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2, 3, 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ διαδικαστικό συμβαστική 8 και έχουμε ένα θέμα διαδικαστικό παρακαλώ Πρόεδρε έχουμε εδώ μια δυσκολία να σας παρακολουθήσουμε, να διαβάζετε και τη σελίδα, γιατί εγώ έχω χάσει τουλάχιστον τρεις-τέσσερις ε, ψήφους. Δεν έχετε διερμηνία. δεν είχα διερμηνία, λέει ο πρόεδρος. Αν μπορείτε να πάτε λίγο πιο αργά, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε επί των τροπολογιών. Okay. Okay. Um, compromise age. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. 6. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 361 και λίμπε 50 Λίμπε 52 τροπολογίες. 361 και Λίμπε 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 51 υπέρ. Κατά. Και πάλι. Ήμκο 51 υπέρ. Κατά. Για να το ελέγξουμε. i Λήξη. Έχουμε έναν ε, από τους σοσιαλιστές που περισσεύει. Και πάλι. Σοσιαλιστές. Εντάξει, λήξη. Εγκρίνεται. Είχαμε την ΙΜΚΟ 51. Μπάτς 10, υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Λήξη. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 363 υπέρ. Κατά. Λοιπόν, καταπίπτει, γιατί δεχτήκαμε την τροπολογία 45, έτσι, η 363 καταπίπτει. Πάμε στην 364, υπέρ, κατά. Για να ελέγξουμε παρακαλώ. Πιθανό να απορρίπτεται. 364. Λήξη. Απορρίπτεται. 365 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 366 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 367 υπέρ κατά για να ελέγξουμε 367 And I close the vote. Λήξη. Rejected. Απορρίπτεται. 368 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 369 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 370 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Γενικό 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Γενικό 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Γενικό 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 371 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 372 υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε. 372. Λήξη. Εγκρίνεται τα 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε. I close the vote. Λήξη. Αγαπητοί συνάδελφοι από τους σοσιαλιστές, δεν σηκώσατε τα χέρια. Δεν μπορώ να ελέγξω λοιπόν. Τι ψηφίζετε. 375 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 375. Λήξη. Rejected. IMCO 56 in favor. IMCO 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. And I close the vote. Accepted. Uh, λοιπόν, 376 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε και πάλι την 376. Λήξη. Απορρίπτεται. 377 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά να ελέγξουμε 48. Πέρας. Απορρίπτεται. 391 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε και πάλι. Την 391. Λήξη. 392 in favor. 392 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 μαζί με την ΕΜΚΟ 61 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μπάτς 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 394 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε. I close the vote. Πέρας. Απορρίπτεται. Μπατ 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μπατ 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 395 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 396 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται.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 Τροπολογία 5.34 υπέρ. Κατά. εποχέ, Απορρίπτεται. σύμβαση 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 549 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο τροπολογίες μαζί. 559 ε, 57 απορρίπτεται 560 υπέρ μετά για να ελέγξουμε 560 And I close. Λήξη. Εγκρίνεται. Είμαι 96 υπέρ. Κατά. Και πάλι. Ήμκο 96 υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε. Λήξη. Εγκρίνεται δύο ταυτόσημες. 563, 564 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 565 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 566 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 567 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήμκο 97 υπέρ κατά για να ελέγξουμε εγκρίνεται λήξεις ψηφοφορίας Κοιτάξτε, εφόσον δεν ε, σηκώνετε τα χέρια σας... Λοιπόν, 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5,70 υπέρ. Λοιπόν, ε, εγκρίθηκε η 83, επομένως θα πρέπει να πάμε απευθείας στη Λίμπε 62. Όλες οι άλλες καταπίπτουν. Λίμπε 62, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 574, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 575 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 576 υπέρ κατά να ελέγξουμε 576 λήξη απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε την 84. Λήξη. Εγκρίνεται. 578 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 585 μαζί με την 586 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται 587 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 588 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 103 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 589 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 590 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 591 μαζί με την ΙΜΚΟ 104 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά εποχές συγκρίνεται δύο τροπολογίες 593 105 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, τρει τροπολογίες, ταυτόσημες 594, 595 και ΙΜΚΟ 106, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται, 596 υπέρ, κατά αποχές Συγκρίνεται, 107 υπέρ, κατά, για να ελέγξουμε, την 107 και λήξη. Απορρίπτεται. Λίμπε 64 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 597 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 598 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 108 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ναι, να ελέγξουμε. Τι είναι 108 ΙΜΚΟ. Λήξη. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές βορύπτεται. ΙΜΚΟ 109 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 600 υπέρ. Κατά. εγκρινεται ελληνικό εγκρίνεται. Υλικό. 1-1-1-111 υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε. I close the vote. Λήξη. Απορρίπτεται. 602 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 604 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 606 υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε γιατί δεν ήταν σαφές για μένα. πλήξη Απορρίπτεται. 607 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 608 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίν, απορρίπτεται 619 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβιβαστική 20α υπέρ κατά για να ελέγξουμε. Συμβαστική 20α ή έλειος 20 bis, λήξη. Απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε και πάλι. Λήξη. Γκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 625 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 626 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 627 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 628 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 629 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6.30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6.31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά Αποχέση εγκρίνεται. είμαι 3 υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 95. Λήξη της ψηφορίας. Απορρίπτεται. 96 um, uh, uh, υπέρ, κατά, αποχές συγκρίνεται. Μπατζένα υπέρ, κατά, αποχές συγκρίνεται. Δύο ταυτόσημες, ΙΜΚΟ 4, Λίμπε, 3 υπέρ. Κατά, αποχές συγκρίνεται. Budget 2 υπέρ κατά αποχές κρίνεται συμβαστική 23 υπέρ, κατά αποχές κρίνεται 103 υπέρ, κατά αποχές κρίνεται 104 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 105 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 106 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 107 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λιμπέ 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 109 υπέρ κατά για να ελέγξουμε την 109 And I close the vote. Λήξη. Απορρίπτεται. Μπάτς 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, απορρίπτεται. Συγγνώμη. 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμικο 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μπάτς 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ. Εποχές εγκρίνεται. 114 and Libe 10. 114 και Libe 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μπάτς 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε 118 λήξη της ψηφορίας εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά Εγκρίνεται. Λίμπε 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβεστή 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβεστή 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 138 πέρας εγκρίνεται 139 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην τροπολογία 7. Γιατί δεχτήκαμε την 138. Περνάμε στην 7. Υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται 141 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 142 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 143 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 147 υπέρ κατά για να ελέγξουμε την 147. Λήξη. Εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 148. And I close the vote. Λήξη. Rejected. Απορρίπτεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 15 υπέρ. Κατά. Ήμκο 15 και πάλι. Υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε. Γιατί δεν ήταν καθόλου σαφές. Λήξη. Εγκρίνεται. 164 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 165 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται 166 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται δήμικο 16 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ήμικο 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήμικο 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται, 69 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 170 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 171 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 171. Να ελέγξουμε. Καλή ιδέα να ελέγχουμε και πού. Λήξη. Απορρίπτεται. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Λίμπε 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε την 181. Λήξη. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά για να ελέγξουμε την 192 λήξη απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 193 υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε οπωσδήποτε αυτή. 193 λήξη. Απορρίπτεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται 195 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 195 λήξη απορρίπτεται 196 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 27 υπέρ κατά Αποχέ απορρίπτεται 197 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία για το σχέδιο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία λήξη συντριπτική πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ψηφίζουμε τώρα την έναρξη των διοργανικών διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 69 γ. Ονομαστική ψηφοφορία επίσης. Άρχεται η ψηφοφορία και λήξη. Συντριπτική πλειοψηφία, συγχαρητήρια στην κυρία εισηγήτρια. Thank ευχαριστώ όλους και ευχαριστούμε και την εισηγήτρια για τη σκληρή της δουλειά αλλά και ολόκληρη την Επιτροπή γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό κυβερνοασφάλεια, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό. Περνάμε. Α, θέλετε το λόγο. Ωραία, εδώ έχουμε λέει κυρία Πιλάρντελ Καστίγιο τελική ψηφοφορία. Τον Οκτώβριο θα γίνει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες για την εξαιρετική συνεργασία. Οι σκιώδεις όλοι ε, και οι βοηθοί βοήθησαν τρομερά. Βεβαίως ήθελα να ευχαριστήσω και το δικό μου βοηθό. Να ευχαριστήσω φυσικά ε, και για την διαρκή ε, βοήθεια της γραμματείας ε, διότι πραγματικά ο, ε, μετά από τόσους διαλόγους, τριμερείς διαλόγους, όλοι στάθηκαν στο ύψος ε, των καταστάσεων. Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι βοήθησαν. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή συγγήτρια. Κοιτάξτε, μετά από κάθε τριμερή αισθάνομαι όλο και καλύτερα. Ναι, Λοιπόν, νομίζω ότι ε, θα πρέπει να δούμε ε, τα πράγματα με πολύ θετική ε, μεριά, ε, ματιά. Ωραία, τώρα είμαστε στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Εδώ ήταν πάρα πολύ δύσκολες και περίπλοκες οι διαπραγματεύσεις. Είχαμε 8 τριμερείς διαλόγους. 8 τριμερείς διαλόγους, οι οποίοι κρατούσαν 3, 4, 5 ώρες ο καθένας. Επομένως, να μην το λησμονούμε αυτό, γιατί διαπραγματευτήκαμε πολλά θέματα και δημοσιονομικά και μερικά είναι πολύ δύσκολα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι. Εδώ είχαμε 8 τριμερίες, πολύ δύσκολες συζητήσεις και επομένως ευχαριστούμε πολύ και την Βουλγαρική Προεδρία που έκανε πάρα πολλά ε, και την προηγούμενη Προεδρία. Τρεις Προεδρίες ενεπλάκησαν στις ε, διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επομένω ψηφίζουμε ε, για την πρώτη συμφωνία ε, βάσει του άρθρου 69F έτσι όπως επιτεύχθη από τις, ε, τους τριμερείς διαλόγους ε, πέρα της ψηφοφορίας ναι, πάρα πολύ ωραία μεγάλη πλειοψηφία, σας ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, στους κοιόδης Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή δουλειά και πολύ καλό το αποτέλεσμα, ενώ δεν ήταν καθόλου εύκολο να επιτευχθεί αυτή η πρόσβαση στο φάσμα ας πούμε το, που είναι θεμελιώδου σημασία όπως γνωρίζετε ε, και όλα τα ε, θέματα που ήταν μέσα σε αυτό το φάκελο ήταν εξίσου σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Ε, πρώτη συμφωνία για τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις, ευρωπαϊκές, για τις ηλεκτρονικές συγγνώμη, επικοινωνίες. Ο κύριος Τοζενόφσκι ε, είναι εισηγητής, έχει και διαδικαστικό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο. Θα ήθελα κι εγώ ε, ε, όπως και η Πιλάρ Δικαστήγιο προηγουμένως ε, να απευθύνω ευχαριστίες στους συναδέλφους, ε, στους σκιώδεις, να ευχαριστήσω και την ίδια την κυρία Πιλάρ Δελκαστήγιο γιατί χρειάστηκε πάντα να έχουμε κάποια συμφωνία αν θέλετε μεταξύ των δύο θεμάτων μας. Να ευχαριστήσω βέβαια και τη Γραμματεία για την τεχνική υποστήριξη και αρρωγή γιατί από τεχνική άποψη αυτό τόσο ο φάκελος ήταν πάρα πολύ δύσκολος γιατί μη ότι η βοηθή χρειάστηκε ε, να ε, συνδέσουν ε, τα δύο θέματα, τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ελεκτρονικών Επικοινωνιών και τον Φορέα Ευρωπαϊκών Εθνιστικών Αρχών για τις Ελεκτρονικές επικοινωνίες. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να επιτύχουμε τεχνικές συμβιβαστικές λύσεις έτσι ώστε να προχωρήσουν τα θέματα και από νομοθετικής απόψεως ε, είχαμε ολονικτίες. Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι μείνανε ξύπνοι μέχρι τις 3 τα ξημερώματα ε, και ευτυχώς ε, είχαμε μια καλή έκβαση. Πιλάρ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθειά σου όσον αφορά αυτήν την ανάγκη παράλληλης αντιμετώπισης των δύο θεμάτων. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και εγώ. Είχατε εξαιρετική συνεργασία. Και τα δύο θέματα ε, έκλεισαν ε, παράλληλα. Δηλαδή στον ε, τριμερή διάλογο ολοκληρώσαμε και τους δύο κανονισμούς. Αυτό ήταν ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την πάρα πολύ καλή δουλειά. Περνάμε λοιπόν τώρα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε λοιπόν για το αποτέλεσμα του ατύπου τριμερούς διαλόγου. Πέρας της ψηφοφορίας. Έχουμε έναν ΕΛΚ ε, παραπάνω. Τώρα είμαστε εντάξει, λέει ο Πρόεδρος. Επομένως, ε, πολύ καλή πλειοψηφία και εδώ. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για μία ακόμα φορά τον εισηγητή και του Σκιώδης. Και περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα που αφορά την ενεργειακή απόδοση. Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας ε, διαδικαστικό από ό,τι βλέπω. Είχαμε δύο εισηγητές. Ε. Στην αρχή είχαμε τον κύριο Γκέρεκ και μετά τον κύριο Μύρος Λαυπόχε. Είμαστε Δημοκρατικό Κοινοβούλιο και επομένως ε, θα δώσω το λόγο και στους δύο εισηγητές εάν τον επιθυμούν. Παρακαλώ, Έντβαρτ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναβληθεί αυτή η ψηφοφορία λόγω του των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς γιατί ε, το κείμενο πρέπει να βελτιωθεί ως προς το περιεχόμενό του και το αιτιολογώ ως εξής το σχέδιο για την ενεργειακή απόδοση ο κανονισμός για την ενεργειακή απόδοση είχαμε ένα συγκεκριμένο στόχο που ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας και ε, άλλο εξοικονόμηση και άλλο απόδοση. Εδώ δεν γίνεται λόγος για την απόδοση, γιατί η εξοικονόμηση ενέργειας δεν ισούται με την ενεργειακή απόδοση, δηλαδή όπου πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμό και να αποδίδεται σημασία στην απόδοση, εκεί υπάρχει η λέξη εξοικονόμηση και αυτά αφορούν τόσο την επικεφαλίδα όσο και το εκτιμώντας 3 και 4 του κειμένου. Για πάρα πολλούς ε, η εξοικονόμηση και η απόδοση ισούνται, είναι ταυτόσιμες έννοιες, αλλά δεν ισχύει αυτό σε επίπεδο φυσικής. Παράδειγμα, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο στόχος η εξοικονόμηση κατά 32% σημαίνει ακριβώς ε, το ίδιο, ότι δηλαδή και ότι η απόδοση θα αυξηθεί κατά 32% μέχρι το 2030. Αυτός δεν είναι ε, στόχος απόδοσης, είναι στόχος εξοικονόμησης. Ίσως ε, όλα αυτά να είναι για κάποιους δύσκολο να τα κατανοήσουν, αλλά η αιτιολογία είναι δύσκολη και οποτεδήποτε λαμβάνουμε μία απόφαση πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις. Η αρνητική χρήση αυτών των όρων και αν ε, τους μπερδεύουμε αυτούς τους όρους αυτό θα σημάνει ότι στην αλυσίδα τροφοδοσίας ε, θα αγνοούνται τα τρία πρώτα βασικά στοιχεία και θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η αγορά. Παρακαλώ πολύ να ε, καταγραφεί αυτό στα πρακτικά. Πολύ ωραία, θα καταγραφεί αυτό στα πρακτικά. Και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Πόχε. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Είναι λίγο δύσκολο για μένα, πώς να σας το πω, να αμφισβητήσω τον κύριο Γκέρεκ γιατί είναι μέρος της ομάδας. Εγώ νομίζω ότι και μεταξύ των εισηγητών, των μελών και μεταξύ των σκιωδών έχει υπάρξει κάποια συνένεση. Ήταν πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσεις, γι' αυτό ευχαριστώ όλους και το προσωπικό το οποίο μας ε, υποστήριξε έτσι ώστε να βρούμε κάποια συμφωνία. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε, ιδεοδός να ψηφίσουμε σήμερα, γιατί εγκρίθηκε το θέμα και από το Συμβούλιο και από την Κομισιόν και από όλους τους ε, ε, σκιώδεις, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Κομισιόν, τον κύριο Νιστόρη, για την σαφή ε, βοήθεια και υποστήριξη στη διάρκεια όλων των τριμερών διαλόγων. Και βεβαίως να ευχαριστήσω, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, ε, την Βουλγαρική Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ κατανοώ ότι αυτή είναι η πρόταση του εισηγητού μας, του κυρίου Πόχε, ε, να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Νομίζω ότι ε, σαφώς ως εισηγητής ε, έχει την έχει την αρμοδιότητα να ζητήσει να γίνει η ψηφοφορία. Βεβαίως, στα πρακτικά θα καταγραφεί η πρόταση του κυρίου Γκέρεκ ως ήθιστε στα πρακτικά της συνεδριάσεως αυτής, οπωσδήποτε θα καταγραφεί το αίτημα του κυρίου Γκέρεκ. Εγώ, Μυροσλάβε, θέλω να σε βοηθήσω γιατί και να σε στηρίξω γιατί αναφέρθηκες ε, στην ε, ε, Επιτροπή. Πραγματικά είχαμε στήριξη τεράστια από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ και το ίδιο ισχύει και για τα επόμενα θέματα. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η ε, στήριξή σας ε, σήμερα. Και οι δύο γενικοί διευθυντές ε, από τις αντίστοιχες γενικές διευθύνσεις και οι ίδιοι οι επίτροποι βοήθησαν να σας πω ότι οι επιτροπές είναι, οι επιτροπές, συγγνώμη, είναι πολύ συχνά παρόντες διαπραγματεύσεις και βοηθούν πολύ τις διαπραγματεύσεις αυτές. Ε, πραγματικά ε, η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, των Επιτρόπων, των Γενικών Διευθυντών, πολύ σημαντική. Επομένω, ενεργειακή απόδοση, ψηφοφορία επί τη προσωρινή συμφωνία προέκυψε από τι διοργανικέ διαπραγματεύσει βάσει του κανόνα 69 F άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Μεγάλη πλειοψηφία και σε αυτή την περίπτωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αποδεχόμαστε λοιπόν το αποτέλεσμα της προσωρινής συμφορίας, συμφωνίας έτσι όπως προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις. Περνάμε τώρα στην προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρόκειται για αναδιατύπωση. Ο Χωσέ Μπλάνκο Λόπες είναι ο εισηγητής μας. Ε, ο κύριος Λόπες. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Πρόεδρο που ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων αλλά αζώντος και εξ ονόματος της ε, Γραμματείας να ευχαριστήσω την Ελβίρα που ήταν πάντα στο πλευρό μας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνεργασία των Κέλλη, Φέντερλη, Ταμπουράνο, Τούρμες που δεν είναι εδώ και την Παλώμα. Να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς τους εισηγητές για την αμοιβαία υποστήριξη. Ταυτόχρονα δε να ευχαριστήσω και τους, τις ομάδες τους και τους βοηθούς τους που μας υποστήριξαν. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και αυτόν που ε, ε, δούλεψε εξ ονόματος της ομάδος μου, τον Αντών και την Πάολα και εξ ε, δικούς μου επίσης τον Επίτροπο Κανιέτε, την ομάδα του και ε, κυρίως στην Πάουλα και τον Αντώνιο, τον Φρανσέσκο και την Άννα Δεχέα. Ε, πιστεύω ότι αυτή η επικοδομητική εργασία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη κρύβεται πίσω από την συμφωνία. Πρόκειται για συμφωνία η οποία μας οδηγεί ε, στην ηγετική θέση όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Δεν έχασε αυτό το ραντεβού στο ιστορικό, το σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι πραγματικά ε, αυτό που είχαμε να κάνουμε το κάναμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ συνάδελφε, λέει ο Πρόεδρος. Ε, θέλετε διαδικαστικό. Ναι, ναι, διαδικαστικό. Έχουμε τόσες ψηφοφορίες. Μήπως θα μπορούσα να ζητήσω με ε, ε, ευγενικά ότι εδώ δεν είναι ομιλίες ε, όταν τους δίνουν το Όσκαρ, ας πούμε, πρέπει να ευχαριστήσουν όλο τον κόσμο. Ευγενικά το λέω, αλλά σας παρακαλώ, μήπως θα μπορούσαμε να επισπεύσουμε λίγο τις διαδικασίες. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ, <clears throat> λέει ο Πρόεδρος. Ναι, αλλά εμείς θεωρούμε ότι ε, αυτά είναι τα προσωπικά μας Όσκαρ. Ε, εμείς σαν να παίρναμε Όσκαρ μιλάμε. Ε, ε, αλλά έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Συμφωνώ μαζί σα. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα. Επομένω, προώθηση χρήση ενέργεια από ανανεώσιμε πηγέ. Περνάμε στην ψηφοφορία. Δεν έχουμε εδώ να δώσουμε άλλα Όσκαρ, ούτε θα ακούσουμε άλλον οσκαρικό λόγο. Ψηφίζουμε λοιπόν για την ε, προσωρινή συμφωνία που προέκυψε από τις διοργανικέ διαπραγματεύσεις βάσει του άρθρου 69F, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Και ε, ολοκληρώθηκε πέρα της ψηφοφορίας. Έχουμε έναν από τη σοσιαλιστική ομάδα παραπάνω, τώρα διορθώθηκε αυτό. Πέρας της ψηφοφορία λοιπόν, μεγάλη πλειοψηφία, 50 ψήφοι υπέρ 7 εναντίον. Εγκρίνεται λοιπόν και περνάμε στο επόμενο θέμα. Ξέρουμε ότι όλες αυτές οι ψηφοφορίες βέβαια ε, θα ε, επαναληφθούν στην Ολομέλη. Αυτό είναι απολύτως προφανές. Αγαπητοί φίλοι, εδώ είχαμε ένα διάλειμμα κατά κάποιο τρόπο στη σκληρή μας εργασία. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ συγκλονιστικά όλα αυτά με αυτές τις προσωρινές συμφωνίες, αλλά εδώ έχουμε μια, ένα ολόκληρο τούβλο με ψηφοφορίες. Ο εισηγητής μας, Γιάκοπ Νταλετούντε, ε, πρόκειται για τους, ε, τα νέα οχήματα πρότυπα επιδόσων για τι εκπομπέ από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Εδώ θα χρειαστούμε πολύ χρόνο. Α ξεκινήσουμε λοιπόν. Συμβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές αποδεκτή. Επόμενη. Ε, συμβασμός ε, με ε, συμβαστική 8. 1-3-2 οι συμβαστικές προτάσεις πρέπει και αυτές να ε, ψηφιστούν υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 10 ονομαστική ψηφορία ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ πρέπει να ε, ελέγξουμε συμβαστική 10 κλείνω την ψηφοφορία γίνεται αποδεκτό, αποδεκτή έτσι λοιπόν ε, προχωράμε τώρα στην ε, τροπολογία 17 και την τροπολογία 18 ψηφίζουμε από κοινού υπέρ παρακαλώ 17 και οι 4 από κοινού υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται 154, 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σε περίπτωση απόρριψης πάμε στο 155 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές αποδεκτό. Αυτή τη φορά γίνεται αποδεκτό. Πάμε στη συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 9. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Η 9. Η εννέα συμβαστική και έκλειση ψηφοφορία. Αποδεκτή. Πάμε τώρα στην 177. 177. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 178 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 179 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 179. Πέρας. Απερίφθη. 180 Απο, ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, δύο τροπολογίες από κοινού, 20 και 182 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Ναι, θέλετε επαλήθευση, παρακαλώ. Δύο τροπολογίες, τροπολογία 20 και τροπολογία 182 από κοινού πέρας της ψηφοφορίας και απερίφθη. Σαν. Ε, τροπολογία 181 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τέσσερις τροπολογίες από κοινού 21, 184, 11, 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται Τροπολογία 185 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα για την 185. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά 185. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Δύο τροπολογίες, 186 και 187 υπέρ. Κατά καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δύο τροπολογίες από κοινού λοιπόν, πέρα της πληροφορία. Απερίφθησαν. Τροπολογία 189 και τροπολογία 190 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Δύο τροπολογίες 191 και 192 από κοινού υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ δεν είναι σαφέ το αποτέλεσμα πέρα τη πληροφορία. και απεριφθήσαν συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δύο τροπολογίες 206 ε, και 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 208 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Επί της 208. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. Τρεις τροπολογίες. Τροπολογία 23, 29 πρώτο τμήμα και τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απεριφθεί. Τέσσερις τροπολογίες. 210, ε, τέσσερις τροπολογίες ε, υπέρ κατά Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Να ελέγξουμε. Πέρασε. Απερίφθη. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 220. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι υπόλοιπε. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh, it was few pages before amendment 153 and 1. Yes, I put it on the list. Good. Yeah. So all of them, uh, six of them fall. Καταπίπτουν έξι τροπολογίες και περνάμε στη 223 υπέρα. Κατά αποχές απορρίπτεται 225 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τη συμβιβαστική 4 υπέρ κατά να, ελέγξουμε να ελέγξουμε ε, την, ε, την συμβιβαστική 4 πέρα της ψηφοφορίας απερίφθη 227 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 229 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 229 και κλείνει η ψηφοφορία. Is rejected. <clears throat> Oh, in favor. 2.30 υπέρ, κατά, ε, πρέπει να προβούμε σε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ηλεκτρονική επαλήθευση του 2.30. Κλείνει λοιπόν η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 2.31 υπέρ. 2.31 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά αποχές ε, μισό λεπτό ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ άρα απορρίπτεται απορρίπτεται 2-3-0 και 2-3-1 είναι ταυτόσιμες και απορρίπτονται 2-3-2 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται Άρα έχετε δίκιο, δεν έπρεπε να ψηφίσουμε στην 231. Τώρα πάμε στην 233. Υπέρ, κατά. Ξανά λοιπόν. 233. Υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 240. Υπέρ, κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ, της 240. και κλείνει η ψηφοφορία. Δεκτή. Δύο τροπολογίες. Υπέρ, κατά, ας το ελέγξουμε. Πέντε τροπολογίες που ψηφίζουμε από κοινού και κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τρεις ε, ε, τροπολογίες. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 2.47 υπέρ, κατά, ηλεκτρονική επανελήθευση παρακαλώ. Η 2.47 Και κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 2.48 υπέρ, κατά, αποχές. Κανείς ε, δεν μπορούσε να αποφασίσει. Δεν σηκώσει το χέρι του. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 2.48. Κλείνει η ψηφοφορία. δεκτή. Ίσως ε, ε, να αλλάξετε χέρι, για μήπως κουράστηκε το ένα χέρι σας. Αλλάξτε με το άλλο και θα είναι πιο εύκολο να ψηφίσετε. Για την επόμενη τουλάχιστον μία ώρα ακόμα. Πάμε στην 2.49. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Υπέρ, κατά, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για την συμβαστική αυτή πρόταση, την 5. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. 2.50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.51 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ. 258. 258. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. 259 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ήτανε οριακά. Η 259 κλείνει ψηφοφορία. Απορρίπτεται απορρίπτεται 2.60 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή 2.67 περίεργη αυτή η κατάσταση και οι 2.68 ψηφίζουμε από κοινού και για τις δύο υπέρ παρακαλώ κατά αποχές ε, δεκτή Συμβαστική 6. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την ηλεκτρονική, ε, για τη συμβαστική 6. Και κλείνει η ψηφοφορία. Δεκτή. Πάμε τώρα στην 269. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Και κλείνει η ψηφοφορία. Δεκτή αυτή τη φορά. Πάμε τώρα στην 271. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.73 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.75 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 27 υπέρ, κατά, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Η 27. Και κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η συμβιβαστική 11 που είναι αρκετά σελίδες πίσω η συμβαστική 11 απορρίφθηκε, ως τούτου καταπίπτει η συμβαστική 12. Και πάμε στην συμβαστική 7 και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ για τη συμβαστική 7. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Ως εκ τούτου 282 υπέρ κατά Παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση. 282 ηλεκτρονική επαλήθευση και κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 284 υπέρ κατά αποχές Νομίζω κανείς δεν θέλει να σηκώσει το χέρι του. Γι' αυτό ηλεκτρονική επαλήθευση. 2.84. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 2.85. Υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 2.85. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 286 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, η ίδια πλειοψηφία απορρίφθηκε και τώρα ε, θα ψηφίσουμε ε, για δύο τροπολογίες, την 287 και την 96 από κοινού, υπέρ, κατά, αποχές, ε, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για αυτές τις δύο τροπολογίες και έκλεισε ψηφοφορία. Δεκτή. Η 28 τώρα. 28 παρακαλώ. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 288 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Η 289 η 2,90 ήταν. Η 2,91 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Οι 30 και 31 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, τα έχω χάσει. Λοιπόν, 32 τώρα ψηφίζουμε γιατί 32 ηλεκτρονικά και έκλειση ψηφορία. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα σε κάποιες τροπολογίες. Για οκτώ θα ψηφίσουμε από την 200 μέχρι την 114. Ε, θα ψηφίσουμε για οκτώ τροπολογίες από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Πάμε τώρα για έξι τροπολογίες από την 33 στην 36 υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτεται. Πάμε τώρα σε πέντε τροπολογίες, αλλά καταπίπτουν όλες αυτές, διότι 154 και 156 απορρίφθηκαν. Πάμε λοιπόν στην 329, 329. Στην επόμενη σελίδα παρακαλώ. 329 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται η 329. 331 υπέρ, κατά, μισό λεπτό, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 331. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Η 331 έγινε δεκτή. Πάμε τώρα κατευθείαν σε, ψηφίζουμε για 7 τροπολογίες. Ε, υπάρχουν 7 τροπολογίες. Από την 355 έως την 365 καταπίπτουν όμως όλες αυτές γιατί οι 154 και 156 απορρίφθηκαν. Η επόμενη τροπολογία για την οποία ψηφίζουμε είναι 362. 362 παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Συγγνώμη γι' αυτό. Η 362 έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίφθηκε η 362. Η 364 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 370 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 374 υπέρ, κατά, αποχές ε, ε, δεκτή. Η 40 υπέρ, κατά. Η 2 υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτεται. Ε, η 42 έγινε δεκτή, η 43-44 από κοινού, υπερκατά, αποχές, ε, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για την 43 και την 44. Δεκτή η 45 υπερκατά αποχές απορρίπτεται, η 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 47 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, η 48 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, η 50 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, η 51, 52, 53 καταπίπτουν. Πάμε στην τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Πάμε στην 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι 61 και 62 καταπίπτουν. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Όχι. Ε, πρέπει να ψηφίσουμε γιατί είναι 61. Λοιπόν, πρέπει να ψηφίσουμε για την 61 και την 62. Λοιπόν, για την 61 ψηφίζουμε για την 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 καταπίπτει, 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 63 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 65 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 71 καταπίπτει, για τον ίδιο λόγο όπως και προηγουμένως, 69 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 70 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, η 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 6 και η 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 74 υπέρ κατά αποχές ε, ας ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 74 παρακαλώ. Και κλείσει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 76 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Η 77 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή η 78 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 80 υπέρ κατά αποχές για την 80. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Λοιπόν, 80 κλείνει η ψηφοφορία. Ναι. Πρέπει να σηκώνετε τα χέρια σας παρακαλώ. 82 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οι 84, 83 και οι 7 καταπίπτουν. Με τα 8, 86, 87 ψηφίζουμε και για τις 3 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Τέσσερις τροπολογίες τώρα. Από την 9 μέχρι την 91. Υπέρ, κατά, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτονται. 93 υπέρ κατά αποχές δεκτή, δεκτές. Πάμε στην 100 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 105 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 4α υπέρ κατά αποχές δεκτή. 118 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για την 118. Κλείνει η ψηφοφορία. Δεκτή η 118. Η 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Διαδικαστικό ο κύριος συγητής πριν από την τελική ψηφοφορία. Κύριε Νταλουντέ, ευχαριστώ πρόεδρε, εκ μέρους των σκιώδων εισηγητών. Θα ήθελα ε, ένα-δύο λεπτά να συζητηθεί το θέμα στην ε, ομάδα γιατί ήταν μια πολύ περίπλοκη ψηφοφορία. Ε, thank you very much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο λεπτά διάλειμμα λοιπόν. Two minutes break. Δύο λεπτά διάλειμμα. Ο συνήθως το κάνουμε αυτό πριν από τελική ψηφοφορία, αν υπάρχει πρόταση από οποιαδήποτε πολιτική ομάδα.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 Final vote. Roll call vote. Jakob Dalunde. Jakob Dalunde για την έκθεση αυτή. Κλείσαμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη ψηφοφορία η συγγήτριά μας είναι η κυρία Ρεμπέκα Χάρμς. Αγαπητοί φίλοι, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Στις 12.30 ε, θα φύγουν οι διερμηνείς ε, και ήθελα να κάνουν και μία δήλωση. Αλλά ε, αν έχει την καλοσύνη γρήγορα, οι διερμηνείς μας τους ακούμε. Οι διερμηνείς ε, διαφωνούν ε, και διαμαρτύρονται για τι ε, επιβεβλημένες συνθήκες εργασίας. Είμαστε επιταγμένοι για αυτή την συνεδρίαση. Ε, Παρ' όλα αυτά, ε, θέλουμε να σα ενημερώσουμε ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση ωραρίου εργασία. Σα ευχαριστούμε πολύ. It means uh, we will finish at 12. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι θα τελειώσουμε ακριβώ στι 12.30. Δεν ε, έχουμε λοιπόν πολύ χρόνο και έχουμε ακόμα πολλέ ψηφοφορίε. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε. Σα ευχαριστώ για τη συνεργασία, κυρία Άρμς. Περνάμε στο θέμα πρόγραμμα έρευνα και εκπαίδευση Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομική Ενέργεια 2019-2020. Περνάμε στην πρώτη τροπολογία υπέρ κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 132 και 133 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε δύο τροπολογίε γιατί ε, αποσύρθηκε 131 Ψηφίζουμε για δύο τροπολογίες. Λήξη. Αγκρίνεται, 137 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές Αγκρίνεται, 135 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. I close the vote. Λήξη. Is rejected. Απορρίπτεται. 134. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 και 140 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 21 υπέρ συγγνώμη και 141 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε 143 λήξη 142 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. 146 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 146. I close the vote. Λήξη. Rejected. Now we vote... Απορρίπτεται. Τμήματική ψηφορία 147 τμήμα 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήμα 2 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε. Τμήμα 2. Ελέγχουμε το τμήμα 2. Close vote. Λήξη. Rejected. 149 in Λοιπόν, 149 υπέρ, κατά. Εποχές, εγκρίνεται. 148 υπέρ, κατά. Εποχές, εγκρίνεται. 150 υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε. Την 150. Λήξη. Εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 153 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 155 υπέρ κατά αποχές ελέγξτε παρακαλώ την 155 λήξη απορρίπτεται 26 και 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 161 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος. Λήξη. Απορρίπτεται. Σαφέστατα. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε. Την 165 λήξη. απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά αποχές. Δεν μπορώ να αποφανθώ να ελέγξουμε την 167. Λήξη. Απορρίπτεται. 168 υπέρ κατά είχε συγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 173 υπέρ κατά για να ελέγξουμε την 173 λήξη απορρίπτεται 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 και 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 176 περ. κατά αποχές εγκρίνεται 31 177 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 και 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 182 υπέρ κατά Αποχές. Για να ελέγξουμε. 182. Λήξη. Εγκρίνεται. Πάμε στις 34. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 185 υπέρ κατά πρέπει να ελέγξουμε την 185 λήξη απορρίπτεται 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 και 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 190 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 41 και 194 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42, 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μαζί με την 196 46 197 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 και 199 υπέρ κατά να ελέγξουμε 49 και 199 λήξη απορρίπτονται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 51 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 202 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε τη 202 Λήξη. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54-204 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 205 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 207 υπέρ κατά Ναι, ελέγξουμε τη 207 λήξη εγκρίνεται 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 209 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 και 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61-211. Ωραία ομάδα. Χάρμ Σταμπουράνο. 61-211 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2-12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 64-65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 68-69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 70 υπέρ κατά για να ελέγξουμε την 70 λήξη απορρίπτεται 71 Τμηματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει το δεύτερο τμήμα. Γιατί οι προηγούμενε τροπολογίες δεν έχουν θετηθεί. Πάμε στην 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ. Κατά άποχε απορρίπτεται 78, λέει ο 76 διορθώνει, υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε, 76. Και λήξη. Απορρίπτεται, 74 υπέρ, κατά. Αποχές. Ψηφίστε παρακαλώ για την 74 λήξη. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε την 79 λήξη. Απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά. Yes, απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Yes, απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 83 υπέρ κατά για να εγκρίνουμε για να ψηφίσουμε συγγνώμη την 83 λήξη απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά εγκρίνεται 88 υπέρ όχι από την 87 πρέπει να περάσουμε στην 89 επειδή εγκρίθηκε κατά πίπτη 88. 89 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Round Ζήτησε να ψηφίσουμε για την 89. Θα πρέπει να ψηφίσουμε την 89. Συμφωνείτε. Αποσύρετε. Δεν το ξέραμε αυτό. Αποσύρετε. Κυρία Μούντι και Μπαλσίτης, αποσύρετε την τροπολογία σας δηλαδή, μάλιστα. Δεν ψηφίζουμε την 89. Την 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Την 90. Λήξη. Απορρίπτεται 91 και 92 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ 94 έλεγχος Υπάρχει έτοιμα ελέγχου της 94 Λήξη απορρίπτεται. Πάμε στην 95 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 7 και 97 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 98 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 8 και 102 μαζί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 9 και 103 μαζί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Δεν ξέρω. Πρέπει να επαναλάβουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 και 108 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τον 10 υπέρ κατά χες απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 και 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 117. Λήξη. Εγκρίνεται. 118 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Την 120. Λήξη. Εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ κατά εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 και 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 και 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ Τι είναι 127 λήξη απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται και τελική ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεσης όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ονομαστική και λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Δεν ήταν εύκολο. Θέλετε κάτι να πείτε. Είστε τόσο ευγενικό πάντα, Γέρζη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα είδο ε, πυρηνική καταστροφή που οργανωστεί για μένα. Όπω I Όπως καταλαβαίνετε, εγώ είμαι ο οργανωτής. Τι μπορούσα να κάνω. η πλειοψηφία αποφάσισε προσεκτικά. Για μένα βέβαια είναι ένα είδο καταστροφής. Θα δούμε βέβαια αργότερα τι θα γίνει με τι εξελίξεις στο θέμα των πυρηνικών. Uh, well, as usual, in the European Union... Συνήθω στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαφωνούμε σε πάρα πολλά σημεία. Αλλά ε, τελικά θα πρέπει να κερδίσει η δημοκρατία. Και εγώ νομίζω, Ρεμπέκα, στην περίπτωση αυτή, πρόκειται περί δημοκρατία. Λυπάμαι. Α υπερασπίσουμε τη δημοκρατία. Το γνωρίζεις πολύ καλά αυτό. Ας πάμε παρακάτω. Έχουμε την έκθεση του κυρίου Κρασνοντέψκη σχετικά με τις υποδομές για εναλλακτικά καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ώρα για δράση. Συμβιβασμικτική ένα υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Όχι, τροπολογία 16 λέει ο πρόεδρος. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Υπέρ, κατά. Αποχές. Θα, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Για την τροπολογία 24. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία διονομαστικής κλίσεω. άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας με μεγάλη πλειοψηφία ε, γίνεται δεκτή. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή, συγχαρητήρια, ευχαριστούμε και τους ε, σκιώδεις. Επόμενη έκθεση του Γιάννη Γκάι. Τροπολογίες ε, για τον Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 19, 2019. Όλοι οι τομεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να τελειώσουμε πριν από τις 12.30 αγαπητοί φίλοι. 201 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.12 υπέρ κατά α, ηλεκτρονική επαλήθευση 2.12 πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη με σαφή πλειοψηφία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 213 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μαζί με τη 214 ταυτόσιμες είναι αυτές 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 215 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 216 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 217 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 218 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 219 και 220 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 221 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 223 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 208 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφοφορία on block από κοινού με οκτώ τροπολογίες από την 76 μέχρι την 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 224 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 225 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 226 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρεις τροπολογίες από κοινού 138 μέχρι 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 227 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τρεις τροπολογίες ε, από κοινού υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνονται. 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω αλλά καλύτερα να υπαλληθεύσουμε παρακαλώ επαλήθευση από τις τροπολογίες 229 πέρας της ψηφοφορίας και απορρίπτεται με μία ψηφοδιάφορα. 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 230 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 231 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 232 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 233 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 197 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα έχουμε block vote υπαριθμών 1 είναι η πρώτη από κοινού ψηφοφορία περίπου 10 τροπολογιών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Block Vote 2. Είναι περισσότερες εδώ οι τροπολογίες. Είναι 10 σελίδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. And now we In favor. 234 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 235 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 236 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 237 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 238 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 239 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 240 μαζί με την προφορική τροπολογία του κυρίου Έλλερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.44 υπέρ κατά Αποχέσε απορρίπτεται 2.45 υπέρ κατά Αποχέσε. καλύτερα να επαληθεύσουμε αγαπητοί φίλοι από τους σοσιαλιστές δεν ψηφίσετε καθόλου. Ο κύριος Τζορίνιο και ο κύριος Ζανονάτο θεώρησαν ότι αφού ψήφισαν στην προηγούμενη ε, περίπτωση δεν χρειάζεται να ψηφίσουν τώρα αλλά είναι σημαντικό θέμα ο προπολογισμό. πρέπει να ψηφίζεται. 2.45 λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 2.45. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Ναι. Και πέρας της ψηφοφορίας και απερίφθη. 2.46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.56 υπέρ κατά κατά απορρίπτεται 2.57 υπέρ 2.57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.60 πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 267 μαζί Α, όχι, χωρίς κανένα άλλο μαζί, καμία τροπολογία. 2,67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 268 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 270 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2,71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2,72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2,73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2,75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τέλεια! Τέλεια, τέλεια. Ε, ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτή την πολύ σοβαρή ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Τώρα έχουμε την κυρία Σοφία Σακοράφα. Ο κανονισμός για γενές διατάξεις του Συμβουλίου υποστηρίζοντας τις τρεθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Τροπολογία 1. Ονομαστική ψηφοφορία. Πολύ σημαντικό η απόρριψη της πρότασης της Κομισιόν. Άρχεται η ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία, πάρα πολύ σημαντικό. Λήξη. Επομένως, απορρίπτεται η πρόταση της Κομισιόν. Τελική ψηφοφορία. Δεν θα ψηφίσουμε τίποτα άλλο στην έκθεση αυτή. Επομένως, ας περάσουμε στα τελευταία δύο θέματα. Um, uh, ο εισηγητή μα, ο κύριο Βιέρινγκ, πρόκειται για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγεία και την τροποποίηση οδηγία. 54 υπέρ, κατά, αποχέ. Ε, Έλεγχο Για την 54 νομίζω ότι απορρίφθηκε. Η 54 παρακαλώ. 54 έκλεισε ψηφοφορία. Δεκτή. Η 55 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Η 56 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Η 57 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Η 58 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Η συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Η 61 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 62 υπέρ κατά αποχές δεκτή 63 υπέρ κατά αποχές δεκτή 64 υπέρ κατά αποχές δεκτή 65 υπέρ κατά έλεγχος 65 έκλειση ψηφοφορία απορρίπτεται η 11 συμβαστική υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 70 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 72 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 12 συμβαστική υπέρ κατά μισό λεπτό ηλεκτρονική επαλήφθηση. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Πάμε στην 79. Υπέρ κατά. Αποχές δεκτή. Η 14 σημαστική, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 83 για την 14 ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για την 14 ε, ηλεκτρονική επαλήθευση, έκλειση ψηφοφορία, δεκτή, με μεγάλη, όχι με μεγάλη, με οριακή πλειοψηφία, αλλά 83 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 84 υπέρ, κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για την 84 84. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 86. Υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Η 16. Συμβαστική υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 17. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 90 υπέρ, κατά, αποχές, απολύπτεται. Η 92, 91 πρώτα απ' όλα, υπέρ, κατά, αποχές, απολύπτεται. Η 92 υπέρ, κατά, απολύπτεται. Η 93 Η 18, η συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Η 97 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Η 19 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Η 101 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 102 υπέρ, κατά, ηλεκτρονική επαλήθευση. η 1.04 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 1.05 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 1.06 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 1.08 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 1.09 υπέρ κατά αποχές δεκτή. ένα ένα ένα υπέρ, κατά, αποχές, επαληθευση ένα επαλήθευση. ένα Και κλείνει η ψηφοφορία. ενα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 115 υπέρ κατά 115 κλείνει η ψηφοφορία Απορρίπτεται. 1-1-6 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτη 117 κατά αποχές ε, δεκτή, η 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 120 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 121 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 122 υπέρ, κατά. ηλεκτρονική επαλήθευση, η 122. Να ελέγξουμε την 122 και κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 123 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ε, η 124 υπέρ κατά αποχές ε, κλείνει η ψηφοφορία για την 124 δεκτή η 125 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24α ε, συμβιβαστική ηλεκτρονική επαλήθευση ε, συμβαστική 24α παρακαλώ ψηφίστε γιατί είναι συμβαστική κλείνει η ψηφοφορία απορρίπτεται πάμε λοιπόν στην συμβαστική 24 υπέρ κατά ε, ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ

Η 1-3-2 υπέρ υπέρ κατά αποχές. Μισό λεπτό πρόεδρε. Η 1-3-2. 2 Πρέπει να σταματήσουμε τώρα. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε χωρίς τους διερμηνείς. Είναι θέμα ε, προάσπισης της ε, δημοκρατίας. Αν συνεχίσουμε μετά τις 12.30 ε, δίνουμε ένα πολύ καλό, κακό με συγχωρείτε, παράδειγμα στην κοινωνία. Εγώ φεύγω. Uh, uh, uh I that still Not... Η ώρα είναι και 29. Δεν είναι και 30. Συγγνώμη κυρία. Μετά από ένα-δύο λεπτά θα μπορούσατε να κάνετε αυτή την παρατήρηση, αλλά όχι τώρα. Μας πήρατε, μας κλέψατε ένα λεπτό. Ε, από τους διερμηνείς ένα μήνυμα. Είναι 36η μέρα των κινητοποιήσεών μας ε, ε, κατά της, μονομερής, της μονομερούς επιβολής άδικων συνθηκών εργασίας για τους διερμηνείς από τη δίκη του Κοινοβουλίου. Λυπούμαστε λοιπόν, να σας ενημερώσουμε, δεν θα δεχτούμε υπέρβαση Εδώ θα σταματήσει η διερμηνία. Uh, citizens' rights, trade union, as you know, is very important for us. So it's just time